ίδιος προσβλέπουμε με μεγάλη αδημονία στις επόμενες συζητήσεις μας του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Ε, η ψηφοφορία θα διεξανθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην σε διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Φερνάντε, πράσινη βίβλο τη Επιτροπή για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λόγο έχει ο εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο στη συζήτηση αυτή που ε, ενεκρίθη με μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με 50 ψήφους, 55 ψήφους υπέρ, 3 κατά και καμία αποχή και Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που με βοήθησαν να φτάσω σε αυτό το σημείο. Τα βιολογικά απόβλητα είναι περίπου το 30% των ανθρωπίνων στερεών αποβλήτων. Είναι εκατομμύρια τόνοι κάθε χρόνο. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι τα απόβλητα αυτά οδηγούν για εκπομπή εκατομμύριων τόνων αερίου αερίων του θερμοκηπίου. Είναι περαιτέρω αέρια θερμοκηπίου από αυτά που εκπέμπονται από τις, ε, την παραγωγή ενέργειας και την αγροτική δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι τα βιολογικά απόβλητα θα πρέπει να περιοριστούν, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να εκμεταλλευτούν οι δυνατότητες που μας δίνουν. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη θέση των αποβλήτων στη συνολική αλυσίδα ανακύκλωση. Χρειαζόμαστε μια νομοθεσία που δεν είναι κατακαιρματισμένη όπως η σημαίνει. Μια νομοθεσία η οποία θα μπορέσει να ξεπεράσει τον κατακαιρματισμό της σε διάφορα νομοθετικά κείμενα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει εναρμόνιση και η κωδικοποίηση αυτής της νομοθεσίας για να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και μεγαλύτερη απλότητα για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ειδική οδηγία για τα βιολογικά απόλυτα για να φέρει νομική ασφάλεια και απλοποίηση ώστε όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς επενδύσεων να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Με το σεβασμό για τις τοπικές ιδιαιτερότητες και για την αρχή της επικορικότητας. Είναι απαραίτητη μια τέτοια οδηγία. Η έκθεση αυτή τονίζει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μείωση των αποβλήτων και μια καλύτερη διαδικασία πρόληψης η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ευρεία τη ενία. Τα καλύτερα απόβλητα είναι αυτά τα οποία δεν υπάρχουν ποτέ. Δεν παράγονται ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη αντιμετώπιση από το δημόσιο τομέα ώστε να αποφύγουμε ότι παραγματικά χάρη οι δημόσιοι κήποι οι οποίοι απαιτούν σημαντική ε, μέρημνα και πάστρα να μην παράγουν ιδιαίτερα απόβλητα ή να χρησιμοποιούνται επιτόπου αυτά τα απόβλητα. Επίσης, η χρησιμοποίηση υπερβολικών συσκευασιών πολλές φορές οδηγεί σε παραγωγή αποβλήτων για τα, τις συσκευασίε για τα τρόφιμα. Γίνεται πολλές φορές μια υπερβολική χρήση στοιχείων στις συσκευασίες. Είναι μεγάλο το πλεονέκτημα για μια κοινωνία της ανακύκλωσης, διότι δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας. Για κάθε χίλιους τόνους ανακυκλωμένων αποβλήτων μπορούν να υπάρχουν 150 θέσεις εργασίας. και όχι απλώς η απόρριψη τους εγωματέρες. Είναι απαραίτητη λοιπόν μια σωστή μέρημνα για τα απόβλητα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, να αντιμετωπίσουμε τη διάβρεση του εδάφους με το να έχουμε μια δυνατότητα αποσύνθεσης σε ευνοϊκές συνθήκες και παραγωγή λιπάσματος από τα βιολογικά απόβλητα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλιστούν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία δημιουργούν πολύ καλά λοιπάσματα και για τη, και για τη γεωργία και μέσω των οποίων μπορεί να υπάρξει μια καινοτομία. Με την προοπτική του 2020, με την προοπτική μια αηφόρου και εφιά ανάπτυξη, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε προ την κατεύθυνση αυτή. Αυτή είναι και η φιλοδοξία τη έκθεση αυτή, η οποία συγχρόνω έχει και ρεαλισμό, θέλει να εξασφαλίσει η επιλεκτική συλλογή των αποβλήτων να γίνει υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους και τις κενότητες, γιατί αυτό είναι σημαντικό και από οικονομική και περιβαλλοντική πτυχή. Γι' αυτό <clears throat> υπάρχει αυτή η φράση στο κείμενο που λέει περνόμαστε φιλόδοξοι και ρεαλιστές συνάμα. Στο Κατσουτιάι, Καλινόφσκι, Κέλλη, Ταμπάτζη, Ολένιακ, Αλφάνο, Γκέρλινγκ, it. Ο κύριος Καλινόφσκι. Ένα λεπτό. Ο κύριος Καλινόφσκι. Mr. Καλινόφσκι, first one minute. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισήγητη. Νομίζω ότι κανονικά δεν θα έπρεπε τα απόβλητα να θεωρούνται πρόβλημα, δεν θα έπρεπε να θεωρούνται ότι μολύνουν την, την, το περιβάλλον. Θα έπρεπε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα υποπροϊόντα των αποβλήτων με χρήσιμο τρόπο και να παράγουμε ενέργεια που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την οικονομική μας ανάπτυξη θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουμε μέσω της ανακύκλωσης τα προβλήματα της ε, υπερθέρμανσης και θα μπορούσαμε να παράγουμε κόμποστ με τον σωστό ευθυνό τρόπο. Αυτό που λείπει είναι οι υποδομές, εφόσον δεν υπάρχουν οι υποδομές Προφανώς δεν προχωράμε και για να υπάρξουν υποδομές απαιτούνται κίνητρα, απαιτούνται χρήματα σε μια πρώτη φάση, χρήματα όμως τα οποία θα βελτιώσουν άμεσα τη ζωή των πολιτών μας, κάτι το οποίο αξίζει. Καταρχήν συγχαίρω τον κύριο Φερνάντες για την έκθεσή του, η οποία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Γιατί οι πολίτες γενικότερα της Ένωσης καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει με τον πλανήτη μας και τις κλιματολογικές αλλαγές και ιδιαίτερα ότι η ατομική συμπεριφορά μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα. Στα σχολεία της χώρας μου όλο και περισσότερο βλέπουμε να, να πετάσουν την πράσινη σημαία και δίνεται πολύ μεγαλύτερη σημασία σε θέματα όπως την ανακύκλωση των αποβιλήτων. Επίσης στον πολιτιστικό τομέα οι γεωργοί καταλαβαίνουν τις αρνητικές συνέπειες των υπερβολικών ποσοτήτων λοιπασμάτων και χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή λιγότερα. Έτσι όλοι μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Και όπως είπαν και άλλοι βουλευτές, όλα αυτά δημιουργούν και νέες θέσεις εργασίας. Ο κύριος Ταμπάντζη. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φερνάντες για την έκθεσή του. Το 2007 θα είχαμε μια άλλη έκθεση για το βιοαέριο που μπορούμε ε, να παράγουμε. Είχα πάρει μέρος στη σύνταξη της έκθεσης αυτής και είμαι ενήμερος για το τι συμβαίνει. Ίσως να έχω και μία μικρά διαφορά με τον εισηγητή εδώ. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έτσι και αλλιώς και τα φυτά και ιδιαίτερα τα ζώα παράγουν αέρια. Και γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξει τις μελέτες και την δυνατότητα, για την δυνατότητα παραγωγής βιοαερίου από την παραγωγή αερίων από ζώα. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι έχουν μιλήσει για άλλα θέματα όπως το κόμποστ, Μιλάμε στην έκθεση Φερνάντες για το του και για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει. Αυτό θα είναι θετικό και από πλευράς περιβαλλοντικής και από πλευράς γεωργικής παραγωγής. Όλα αυτά είναι σημαντικά βήματα που μπορούμε να πάρουμε με ευθυνό σχετικά τρόπο. Έχουμε σε ορισμένες περιοχές ειδικά χαρακτηριστικά και ειδικά προβλήματα είτε για την βιομάζα, είτε για τα βιοαέρια, είτε για το κομπόστ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συνενώσω τη φωνή μου με αυτή των προλαλισσάντων που εξέφρασαν συγχαρητήρια προς τον εισηγητή κ. Φερνάντζ. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα διότι η προβληματική του διαχωρισμού των αποβλήτων μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε κάνει αρκετά. Χωρίς τη σωστή διαδικασία διαχωρισμού δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα βιοαπόβλητα με το σωστό τρόπο. Υπάρχουν όμως τόσες πολλές δυνατότητες ενώπιόν μας. Οι εγκαταστάσεις βιο... φυσικού βιοαερίου χάρη, που θα πρέπει να υποστηριχθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται υποστήριξη των διαρθωτικών ταμείων σε περιφερειακό επίπεδο, επίσης και σε επίπεδο τοπικό. Μπορεί να δημιουργηθεί παραγωγή ηλεκτρισμού παραγωγή χάρη από το βιοαέριο που θα είναι πιο ε, αποτελεσματική αυτή η διαδικασία. Κύριε Φάλλο για ένα λεπτό. Κυρία Φάλλο. Είναι μια πολύ καλή έκθεση και το συγχαίρω. Με έχει εντυπωσιάσει μία από τις πρώτες φράσεις της αιτιολογικής έκθεσης. Λέγει συγκεκριμένα ότι η πολιτική διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να οδηγήσει στη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κοινωνία ανακύκλωσης. Υπάρχουν αντιφάσεις βέβαια σχετικά με τη διαφοροποίηση των αποβλήτων και κατά πόσον θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και όχι μόνο οικολογικά αλλά και οικονομικά. Πολλές φορές τα διάφορα κράτη μεταφράζουν με τον δικό τους τρόπο τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Δεν πρέπει λοιπόν να περιοριστεί σε συμβολές η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φιλόδοξες και αποφασιστικές απαντήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην κρυβόμαστε πίσω από το μέγεθος των προβλημάτων. Οι στόχοι είναι επιτεύξιμοι. Ας ακολουθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Ξέρουμε ότι έχουν περάσει σε ειδικά μέτρα ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Έχουν διαβάσει την έκθεση αυτή, τη βρίσκω ότι είναι απόλυτα πλήρης και περιεκτική για όλα τα θέματα τα οποία συνδέονται με τα δύο απόβλητα, χώματερε, απώλεια ενεργειακών πόρων, ανάγκη ε, ποιότητος, κομποστοποίηση κτλ. Με μεγάλη λύπη πρέπει να πω ότι έχω διαφωνία με τον κύριο Φερνάντες. Δεν τον παρακολουθώ στο σημείο όπου αναφέρεται σε υποχρεωτικό, υποχρεωτικό διαχωρισμό στη συλλογή αποβλήτων. Αυτό το αρνούμε επί της βάσης της επικουρικότητας και Διαφωνώ γιατί προσπαθεί να παγιώσει μια μέθοδο η οποία έχει ξεπεραστεί σε πολλά μέρη από μεθόδου υψηλή τεχνολογία για τη διαφοροποίηση των αποβλήτων. Είναι πεπαλαιωμένη αυτή η μέθοδο μέχρι πρωτού καν την εφαρμόσουμε. Αυτό θέτει την ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο χειρότερο δυνατό επίπεδο. Δεν δέχομαι να ζητήσουμε περαιτέρω ρύθμιση αντί να προτείνουμε περαιτέρω κίνητρα και ζητώ από την Κομισιόν να αρνηθεί αυτή την έκκληση για υποχρεωτική διαλογή των αποβλήτων. Αναφέρθηκα στα ονόματα κύριε Μπόρις για να είναι σαφές ότι αν κάποιος δεν είχε αναφερθεί το όνομά του θα έπρεπε να ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, επειδή παραμένετε εδώ πέρα και ξενυχτάτε όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, σα δίνω το λόγο. Αλλά λέω τα ονόματα των συναδέλφων στην αρχή, αν δεν έχει ακουστεί το όνομά σα πρέπει να διεκδικήσετε και να λάβετε το λόγο. Κύριε Μπόρι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τη γενναιοδορία σας και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεση του το 30% των αποβλήτων μπορούν να ανακυκλωθούν. Δεν ξέρω αν έχουμε βέβαια όλοι τις κατάλληλες δομές για την ανακύκλωση γιατί οι περισσότερες χώρες της Ανακεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης δεν διαθέτουν τέτοιου είδους υποδομές. Πρέπει λοιπόν να τις βοηθήσουμε διότι αυτό είναι ο λογικότερος τρόπος να χειριστούμε τα βιοαπόβλητα και είναι σωστό να προσπαθήσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή ενέργειας. Η Δανία είναι υπόδειγμα διότι εκεί υπάρχουν οι υποδομές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα πρέπει να γενικευτεί και να το αναφέρουν και οι δημοσιονομικές προοπτικές του μέλλοντος. Επιτροπής και του Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και για αυτή την έκθεση, αυτή τη φορά για τα βιοαπόβλητα. Και ευχαριστώ και τα μέλη του Κοινοβουλίου που εξέφρασαν τις απόψεις τους και αποτελούν πολύτιμη συμβολή στη συζήτηση. Όπως θα ξέρετε, στις 18 Μαΐου η Κομισιόν ενέκρινε μια δήλωση, ανακοίνωση για τα μελλοντικά βήματα της ανακύκλωσης των βιοαποβλήτων στην Ένωση που συνοδευόταν και από μια προσθήκη με συγκεκριμένες λεπτομερείς τεχνικές αναλύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό της και σε κάθε μία από τις χώρες που την αποτελούν οι υπηρεσίες μας παρακολούθησαν όλες τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο για τα βιοαπόβλητα και βρίσκω πολύ ενθαρρυντικό ότι καταλήξαμε στα ίδια γενικά συμπεράσματα ότι υπάρχει δηλαδή βέβαια χώρος για βελτίωση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων και ότι η βελτίωση αυτή μπορεί να αποφέρει και θετικά οικονομικά και περιβαλλοντολογικά αποτελέσματα. και όλα αυτά φυσικά θα συμπληρωθούν και από νομοθεσία όπως η οδηγία για τα σχωματεράς. Εδώ πρέπει να εφαρμοστεί βέβαια και η αρχή της επικουρικότητας. Η βασική διαφορά μεταξύ της δικής μας προσέγγισης και του εισηγητή αφορά το θέμα μιας πιθανής μελλοντικής οδηγίας για τα βιοαπόβλητα. Εμείς δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται μια τέτοια χωριστή οδηγία γιατί η διαχείριση μπορεί να βελτιωθεί με καλύτερη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και γι' αυτό θα αναλάβουμε ορισμένα προγράμματα διαχείρισης των βιοαποβλήτων και καθορισμό κριτηρίων ε, για την ποιότητά τους και την ποιότητα της ανακύκλωσης και την καλύτερη χρήση τους. Καθορισμό δηλαδή ελαχίστων κριτηρίων μετά την αναθεώρηση και των σχετικών οδηγιών και τον καθορισμό στόχων για τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων. Τουλάχιστον το 2014 θα έχουν γίνει όλα αυτά. Ολόκληρη δέσμη προτάσεων δηλαδή και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είστε διατεθειμένοι να μας υποστηρίξετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο σημερινή σε διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Ολένια η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και ο ρόλος των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική